Good morning, everyone. Thank you for uh, coming. If there are no objections, uh, the agenda for today. Καλημέρα σας. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ένα workshop για τη ρομποτική στην ε, δημόσια υγεία με την Σολεδά και τον Λουίς που το οργανώνουν αναμένεται για την 3η 19 Φεβρουαρίου από τις 3 και μετά και σας περιμένουμε. Έχουμε σήμερα 16 γλώσσες διερμηνία και μετάδοση στο διαδίκτυο με web streaming της συνεδρίασης. Έχετε επίσης τα πρακτικά της συνεδρίας 16ης της 6ης Δεκεμβρίου του 2018 δεν έχετε αντίρρηση. Εγκρίνονται τα πρακτικά και σας ενημερώνω για τις δύο οργανικές διαπραγματεύσεις ε, για την προαγωγή καθαρής και αποτελεσματικής ενέργειας ε, στα οχήματα που κινούνται στις οδικές μεταφορές. Έχει εξασφαλιστεί συμφωνία σε σχέση με θέματα που έχουν να κάνουν και με τις υπηρεσίες και με την ρήτρα αναθεώρηση, αυτά δηλαδή που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο για την περίοδο μετά το 2030 και τους στόχους. Επίσης, αποκλείονται όπως είχε ζητηθεί οι παραπομπές στα βιοκαύσιμα και οι στόχοι. Και επίσης υπάρχει και δυνατότητα το Κοινοβούλιο να επανέλθει προκειμένου να επιτύχει ε, φιλόδοξους στόχους το 2030 τόσο όσο και στην προηγούμενη περίοδο. Επίσης για τα τρόφιμα, νομοθεσία, γενικός, γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, καλή μέρα η Δευτέρα όπως βλέπετε, συμφωνία και εκεί. για το χρόνο της δημοσίευσης τη διαχείριση, την διαγραφή καλύτερα των, δικαιωμάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων και τον κατάλογο των εμπιστευτικών θεμάτων, ε, όπως ενσωματώθηκε δηλαδή η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια δυνατότητα για ε, προσφυγή με το άρθρο 61, εξάμεινη ε, περίοδος επιβολής ποινικών ρητρών, κοινοποιήσεις και ολοκλήρωση ε, των αυτοψιών ε, μέσα σε τετραετία. Αυτό λοιπόν ψηφίζεται στην Επιτροπή μας στις 20 Φεβρουαρίου, το General Food Law. Και η πρώτη δεν την ανέφερα, η προηγούμενη με την ε, με τις καθαρές και αποτελεσματικές ε, τεχνολογίες στα καύσιμα, 27 Φεβρουαρίου ψηφοφορία. Διοξίδιο του άνθρακα εκπομπές, τρίτος άτυπος τριμερής διάλογος. Συζητήθηκαν τα έκρεμη ζητήματα χωρίς να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις. Λιγότερο πολιτικού χαρακτήρα ζητήματα όπως το πλαίσιο προαγωγής, η ενημέρωση του ΑΠ, του ΒΕΚΤΟ, το pooling, ε, συνθετικές, τα συνθετικά καύσιμα, προηγμένα καύσιμα έχουν προσωρινά συμφωνηθεί. Ενώ οι συζητήσει για τα EMS στο επίπεδο ε, της ε, υπέρβασης και των ΣΛΕΒ θα συζητηθούν στον προσεχή τριμερή διάλογο την επόμενη εβδομάδα. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία μας. Έχετε πιστεύω την, ε, το πάκο με, τους, ε, με τις ψηφοφορίες. Ο κύριος Λαβία είναι ο υπέτειος. Θέλετε το λόγο κύριε Λαβία. Πρόεδρε ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου ξεκινώντας να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ηγητές. Πριν να ξεκινήσει κατάλογο, πριν κατα... ξεκινήσει η ψηφοφορία, μεγάλη δουλειά κάναμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ τη γραμματεία, ευχαριστώ το προσωπικό των πολιτικών ομάδων για, και βέβαια και το δικό μου το προσωπικό για όσα έκαναν τις τελευταίες εβδομάδες που ε, μέρα και νύχτα δούλεψαν για να ε, καταστήσουν δυνατή την σημερινή ψηφοφορία. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να τους ευχαριστήσω όλους. 1.300 από τις 2.000 τροπολογίες που είχαν κατατεθεί έχουν καλευθεί από τις συμβιβαστικέ. Τεράστια προσπάθεια σας διαβεβαιώ. Όλοι όμως ε, συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου με τη συνεργασία της τους. Λυπούμε που θα σας ε, ταλαιπωρήσω με ένα μακροσκελή κατάλογο ψηφοφοριών σήμερα. Είναι όμως θέμα πολύ περίπλοκο αυτό και είναι η πρώτη φορά που έχουμε αρμοδιότητα συνομοθετική με βάση το άρθρο 54 με την Επιτροπή Άγκρη, εμείς η Επιτροπή του Περιβάλλοντος, για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα και έτσι είναι απαραίτητο να γίνει η ψηφοφορία μας μέσα στα χρονικά πλαίσια έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε το θέμα ολοκληρωμένο με τη δική μας θέση μέσα στην Ολομέλεια Εγκαίρο. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλά αποτελέσματα στην ψηφοφορία. Η πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αρχίζουμε. 241 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές και επαληθεύουμε. Αρχίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 242 υπέρ. Κατά. Αποχές επαληθεύουμε 242. Πέρας. Απερίφθη. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 244 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Πέρας. Και απερίφθη. ...245 υπέρ... ...κατά... ...άποχες... ...επαληθεύουμε... ...ναι, είναι καινούρια η αίθουσα αυτή που χρησιμοποιούμε πρώτη φορά... ...πέρας... ...εγκρίνεται... 246 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 247 υπέρ, κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Η πράσινη ήταν μοιρασμένη σε αυτό. Ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν. 248 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη. Βλέπετε όμως το αποτέλεσμα. Ίσα ίσα. 251-252 ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές επερίφθησαν. 254-255 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται εγκρίνεται 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 258 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 287 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 9 τώρα παρακαλώ. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 337 υπέρ σελίδα 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται people if they are still arriving, because then I will have to start checking because it's too close. Compromise 3, who is in favor? Συμβαστική 3, παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 19. 400 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Σελής 23, τροπολογία 434, υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 4, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 453 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 454 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε 454 πέρας και εγκρίνεται 456 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 455 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 457 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 458 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 459 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 460 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 461 υπέρ κατά Αποχέ απερίφθη 462 υπέρ κατά αποχέ απερίφθη 463 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 464 υπέρ κατά αποχέ απερίφθη 465 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5β υπέρ Κατά. Επαληθεύσουμε παρακαλώ είναι και συμβαστική. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σελής 32. «523. Υπέρ. Κατά. Αποχές επερευθεί. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 573 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική 9 β υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σελίδα 41. 630 Υπέρ. Κατά. Αποχές Ας επαληθεύσουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 631 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 632 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 634 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 635 υπέρ κατά, εποχές, επαληθεύουμε. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 636 υπέρ. Κατά. Ποχές. Κύριε Τσάλτερς. Επαληθεύουμε. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 637-638 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 640 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 643 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 654 υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. 655 υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. 656 υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. 657 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 658 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 659 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 660 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 661 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 662 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 663 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 664 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 665 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 666 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 667 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 668 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, παληθεύουμε. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται πράγματι. Συμβαστική 11. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 684 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 685 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 686 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 687 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 688 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 689 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 690 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 691 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 692 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 693 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σελίδα 56. Τροπολογία 804 υπέρ. 804. Σελίδα 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαληθεύουμε. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 812 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα. I'm 814. 814 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 815 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 816 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 817 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 818 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 819 υπέρ κατά εποχές ας επαληθεύσουμε. Still, eight, uh, still 59, It's closed. Λήξη σοφορίας εγκρίνεται. 821. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται 823 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται 820 μ, όχι 825 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 827 υπέρ κατά Εποχές επαληθεύουμε. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 828. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 829. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 830 υπέρ. Να, καταπίπτει. Οκτώ τριάντα υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 8.32 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 8.34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8.39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8.40 block vote υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 841 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 842 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 843 υπέρ. Κατά. εποχές Επαληθεύουμε. Closed. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 870 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 871 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 872 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 873 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 915 υπέρ. Είμαστε στη σελίδα 64. Τροπολογία 915 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16α υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε. The vote is open and the vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περάμε σελίδα 66, τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 9.32 υπέρ. Κατά. Εποχές. Επαληθεύουμε. Την 9.32. The vote is uh, close. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 9.33 υπέρ. Κατά. Μπορείτε παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σε 9.33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε. It was a delay in hands, I must say. It's closed. Λήξη. Εγκρίνεται. 9.34 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 9.37 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 9.38 υπέρ. Κατά. εποχές ε, παληθεύουμε. Κύριε Έκχαουτ, ψηφίζετε κατά της ίδιας σας τροπολογίας. Ψηφίσατε, κατά. Με έχετε μπερδέψει. Λήξη, λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 9.39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9.40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επαληθεύουμε. 9.40. And Λήξη ουσφορίας. Απορρίπτεται. 941 υπέρ. Κατά. Εποχές. Παληθεύουμε. Λήξη. Εγκρίνεται. 9.43 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 9.44 υπέρ κατά, εποχές. ας επαληθεύσουμε. Παρακαλώ, μην ψηφίζετε και ναι και όχι. Σηκώνετε το χέρι σας και στις δύο περιπτώσεις. Εγκρίνεται 9.45 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 9.46 υπέρ. Κατά εποχές Επαληθεύουμε. Την 946. Λήξη. Απορρίπτεται. 947 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 948 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. 9.48 Λήξη. Εγκρίνεται. 949 υπέρ. Κατά. Εποχές. Γκουε τι κάνει. Υπέρ. Εγκρίνεται. 950 υπέρ. Κατά. Εποχές. Επαληθεύουμε. έχουμε και ένα νέο παίκτη. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 9.51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9.52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Λήξη ψηφοφορία Εγκρίνεται. 9.53 και 9.54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτονται. 9.55 υπέρ κατά, εποχές, απορρίπτεται. 9.56 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 9.57 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 9.58 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 9.60 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 9.61 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 9.62 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε. Λήξη. Εγκρίνεται. 9.63 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά, εποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 969 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 970 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 9 Συμβαστική 18β υπέρ, κατά, εποχές, επαληθεύουμε. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 9.58. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εποχές. Επαληθεύουμε. Την 9.85. Λήξη τη Απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Ε, μια ομάδα που ξεκινάει από τη 1246. Ποιος είναι υπέρ. Σελίδα 71 είναι ένα μπλοκ τροπολογιών που ψηφίζονται όλες μαζί ξεκινάμε, ξεκινάνε από τη 1246 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Λήξη. Απορριπτώνται. Συμβαστική 19β υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε σε 76. Τροπολογία 1032. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Απορρίπτεται. 1033. Υπέρ. Κατά. Α Ας επαληθεύσουμε. Απορρίπτεται. 10.35 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 10.36 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 1037 υπέρ. Κατά. Να σε παληθέψουμε. Λήξη της Απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10.47 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Πρέπει σελίδα 84. Δέκα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11.20. 1120 υπέρ. Κατά. Εποχές. Ας επαληθεύσουμε. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11-21 Υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 11-22 υπέρ. Κατά εποχές επαληθεύουμε. Λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται. 11-23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Σελίδα 92 1199 υπέρ. Κατά. Εποχές. Ας επαληθεύσουμε. 1199. απορρίπτεται. 1200 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 1201 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σε επόμενη σελίδα. 1240 1238 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 1240 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 1239 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 1242 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 1241 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 1244 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 1243 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται 1245 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 1247 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 1248 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται 1249 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται 1250 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1251 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1253 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1254 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτεται. 12.55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12.56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12.57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12.58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12.59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12.60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ 62 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τη 1263. Τέλος, απορρίπτεται. 26 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είμαστε στη σελίδα 100. 1285 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103, σελίδα. 27 συμβεβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 σελίδα, 1337 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1338 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1349 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1350 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1351 και 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1355 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1354 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1355 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1365 1365 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, επαληθεύουμε παρόλα αυτά. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε τη 1365, παρακαλώ πολύ ψηφίστε. Εγκρίνεται. Δεν νομίζω όμως ότι ψήφισαν όλοι. Δεν μπορούσα να το προβλέψω αυτό το αποτέλεσμα. 1372 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1373 απορρίπτεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ. Κατά επαλήθευση. Συμβιβαστική 30. Κυρία Ντάλη, δείχνατε κατά. 30. <clears throat> Εγκρίνεται. 112 δώδεκα σελίδα. 14.03 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14.04 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 14.05 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14.06 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14.07 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14.08 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14, 13 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Έλεγχος 14, 13. Νομίζω ότι ένας επιπλέον ψήφισε από τους σοσιαλιστές. Κάποιος πρέπει να βγάλει την κάρτα του από τους σοσιαλιστές. Εντάξει. Μάλλον παραπάνω που ένας βγάλατε την κάρτα σας. Τέλος. Απορρίπτεται. Κάπως πρέπει να το ρυθμίσετε αυτό, γιατί υπάρχει σύγχυση. Χρειάζεται κάποια καθοδήγηση. Προσπαθώ να το κάνω, αλλά δεν είναι και δικιά μου δουλειά. Να επαναλάβουμε την ε, ψήφο, γιατί στους σοσιαλιστές επικρατεί σύγχυση. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για το 14-13. Πέρας εγκρίνεται. Δεκατέσσερα, δεκατέσσερα, υπέρ. Κατά, αποχές, ελέγχουμε. Πέρας, απορρίπτεται. 17.95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η δεν ψηφίζεται. Εντάξει. Επαληθεύουμε λοιπόν την 1495. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 14-15 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14-24 υπέρ, κατά, αποχές, 1441 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14-16 υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε. Τέλος, εγκρίνεται. 31 συμβιβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14-23 υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε. 23, 14, 23. Τέλος. Εγκρίνεται. 562 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε. Αρχή της ψηφοφορίας, τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. υπέρ. Κατά αποχές 1426 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1427 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1428 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1429 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1430 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1432 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1431 υπέρ κατά, αποχές, επαληθεύουμε την 1431. Αρχή της ψηφοφορίας, τέλος, εγκρίνεται. 1433 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1434 υπέρ, κατά, αποχές, Επαληθεύουμε. Συμφωνούν όλοι. Α, όχι, εγκρίνεται. Δεκατέσσερα τριάντα πέρα. Κατά αποχές. Επαληθεύουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 1436 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πλειοψηφία. Υπέρ μάλλον, αλλά ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Με την ίδια πλειοψηφία. Απορρίπτεται. 1437. Κατά αποχές απορρίπτεται. Α, συμφωνούν όλοι για αυτήν την τροπολογία, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, εγκρίνεται. 14.38. Υπέρ, όλοι, κατά. Απορρίπτεται. Επαληθεύουμε τη 14.38. Πέρας. 29. Απορρίπτεται πάντως. 14.39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14.40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14.42 κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14.43 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14.44 υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε. Αρχή της ψηφοφορίας, τέλος. Απορρίπτεται. 14.45 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 14.46 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 14.47 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14.50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14.51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14.52 και 53 υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε. Τέλος εγκρίνεται. 1454 καταπίπτει, 1455 υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε. Αρχή της ψηφοφορίας, τέλος, εγκρίνεται. 1456 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14.57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14.58 υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε. Πέρας, απορρίπτεται. 14.59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14.60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1461 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1462 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1463 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1464 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1465 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1466 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1467 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1471 υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε. 1471 Πέρας. Απορρίπτεται. 1472 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1473 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1474 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1475 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1476 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1478 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1477 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1480 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1479 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1481 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1483 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1482 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1484 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1485 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1487 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1486 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1488 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1489 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1490 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1491 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1492 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. 1492 αρχή της ψηφοφορίας Πέρας. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14.93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14.94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14.95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1496 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1497 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1498 υπέρ κατά επαληθεύουμε 1498 πέρας Εγκρίνεται. 1500 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1501 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές 1515 15-15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15-14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 15-16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15-17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15-18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15-19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15-20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15, 21, 22, 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15, 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25, 26, 27 και 28 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 15, 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφτεται. 15, 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφτεται. 15, 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφτεται. 15, 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, ελέγχουμε τη 1532 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίψετε. 1533 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. 1534 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίψετε. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15.35 υπέρ κατά ελέγχουμε. 15.35 Τέλος απορρίπτεται. 15.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αυτή είναι καλή συμβιβαστική. 134 σελίδα. Συμβιβαστική 48. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. 1693 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1694 υπέρ. Κατά αποχές 1715 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επαληθεύουμε. Αρχή της ψηφοφοριας 1715. 17-15. Τέλος. Απορρίπτεται. 17-16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 143 σελίδα. Ψηφέσουμε την 1793 ε, υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 1794 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Όχι. Έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη. 49 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1796 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση. 1796. Τέλος. Απορρίπτεται. 6.33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15.02 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 συμβιβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ, Ναι, δεν ήταν σαφές να ελέγξουμε το αποτέλεσμα της 65. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Παρακαλώ πολύ σηκώνετε τα χέρια σας. 66 υπέρ. Κατά επαλήθευση. 66. Τέλος. Εγκρίνεται 66. 67 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. It's closed. Εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 70 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 72 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 73 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 74 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 75 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε αρχίζουμε πέρας και απερίφθη 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ. Κατά. Αποχές επαληθεύουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 78 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη. 92 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 95 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 96 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη. Εκατό. Υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 35 υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 100... Συμδιορθώνει Πρόεδρος. Συμβαστική 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 110. Τροπολογία 110 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 ε, υπέρ. Κατά Αποχές, η πράσινη είναι υπέρ. Εσείς απέχετε. Ας το επαληθεύσουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 115 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 116 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 117 υπέρ κατά επαληθεύουμε Πέρας. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 129 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη, συμβαστική 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη. 145 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 146 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί ε, με μεγάλη πλειοψηφία επελθεύουμε όμως πέρας απερίφθη 147 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 150 υπέρ. 149. Επεληθεύουμε βεβαίως. Αρχίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Αλλάξατε όμως πλειοψηφίες ε, στις ψηφοφορίες του κύριου Φλάνναγκαν, στο απολογίες του κύριου Φλάνναγκαν. Δύσκολο λοιπόν να μην μπερδευτεί κανείς. 150 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές, απερίφθη. 151 υπέρ κατά... Ας επελθεύσουμε. πέρας και απερίφθη. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 155 υπέρ κατά, αποχές και επαληθεύουμε. And it's closed. And it's rejected. Πέρασε περίφθη 40 συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. απερίφθη, 164 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 165 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 166 υπέρ. Κατά αποχές υπερήφθη. 167 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 168 υπέρ. Κατά επαληθεύουμε. 168 πέρας απερίφθη 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 171 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 186 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 180 έστω 192 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 193 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 194 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 195 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 196 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 συμβαστική υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 6 υπέρ κατά επαληθεύουμε. Αρχίζουμε και πέρας. Και απερίφθη. 202 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 44 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 210 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 210 υπέρ κατά αποχές απερίφθη να επαληθεύσουμε τη 211 Πέρας. Εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 219 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 220 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 221 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 222 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 223 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε 223 Μα πού είναι αυτός ο κύριος Φλάναγκαν. Τόση πολύ ταραχή που έχει προξενήσει. Πέρας. Να, τα. Τα βλέπετε. Απερίφθη. Διακόσια 224. Ας πάμε κατευθείαν στον έλεγχο. Γιατί άλλαξαν οι ισορροπίες. Πέρασε. Απερίφθη. 225, 226, 227 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ΕΛΚ τι είναι υπέρ κατά. Υπέρ. Εγκρίνεται. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ. Επαληθεύουμε. ...229 πέρας και εγκρίνεται αυτή τη φορά. 230 υπέρ. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 231 υπέρ. Κατά Αποχές απερίφθη 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ. Συμβαστική 46 εγκρίνεται. 236-237 υπέρ. Κατά Αποχές απερίφθησαν 238 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 239 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 240 υπέρ κατά αποχές απερίφθη και επαληθεύουμε βεβαίως τη 240 Πέρας. Και εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ θερμά για την επαλήθευση και εννέα υπέρ κατά απερίφθη θα έλεγα αλλά ας επαληθεύσουμε την εννέα. Πέρας, απερίφθη. Και να τα τελειώσαμε τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ η γραμματεία να επαληθεύσει αν υπάρχει δυνατότητα για διόρθωση στην 1120 σελίδα 24, 84. Σα είπε η γραμματεία ότι έπρεπε να έχει ψηφιστεί, αλλά εγώ νομίζω δεν έπρεπε να έχει ψηφιστεί. Μας ξέφυγε κάτι? Uh, Μα δεν έπρεπε να ψηφιστεί, γιατί είχαμε ήδη εγκρίνει άλλη προηγουμένω και καταπέσει. Καλώ. Εντάξει, υπερψηφίσαμε που λένε, παραψηφίσαμε. Μία παραπανήσια που έπρεπε να έχει καταπέσει. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζουμε. And εγκρίνεται και συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν πάνω στο φάκελο, τον κύριο αλλά και τους λοιπούς. Ολοκληρώνουμε έτσι τη σημερινή μας συνεδρίαση. Ένα λεπτό, ακούστε με λίγο. Θα σας ενημερώσω λοιπόν ότι η συνεδρίασης που είχε προβλεφθεί για τις 21 Φεβρουαρίου, 21 Φεβρουαρίου έχει ματαιωθεί. Μην έρθετε, κατά λάθος.